przewodniczący! Παρακαλώ λάβετε τις θέσεις σας. Θα αρχίσουμε λοιπόν την πρώτη ε, ώρα των ερωτήσεων σε λίγα λεπτά. Otwieram posiedzenie. Protokół wczorajszego posiedzenia. Ε, τα πρακτικά της εξήνή συνεδριάσεως και άλλα έγγραφα είναι διαθέσιμα, ε, οπότε θέλω να ακούσω αν έχετε παρατηρήσει επ' αυτού. Δεν ακούω κάτι τέτοιο, οπότε ε,